Γεια σας, συνεχίζουμε την εργασία μα. Σήμερα το πρωί, καλύτερα, είχαμε πολλές συζητήσεις. Και σήμερα το απόγευμα έχουμε μια σειρά από ψηφοφορίες και προτού περάσουμε σε μια εργόδη διαδικασία ψηφοφορίας και έρχονται βουλευτές έτοιμοι με τις κάρτες αναχείρε. Ας χρησιμοποιήσουμε αυτή την ώρα για να αναφερθούμε στα θέματα της διαφθοράς. Για πρώτη φορά στη θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της ε, τρέχουσας θητείας τουλάχιστον, έχουμε ξεκινήσει με το θέμα της διαφθοράς, το οποίο βρίσκεται σε υψηλό σημείο στην ημερήσια διατάξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και της Κομισιόν. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ θετικά. Αγωνιζόμαστε εναντίον της διαφθοράς. Προσπαθούμε να θεσπίσουμε ευρωπαϊκά πρότυπα σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο αναλύουμε την κατάσταση και προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το μεγάλο κακό. Αυτή τη μάστιγα κατά της ε, ευρωπαϊκής αλλά και κατά των πολιτών που στρέφεται εναντίον των θεσμών των Εθνικών αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πολύ καλό λοιπόν το ότι η Κομισιόν μας έχει δώσει μια έκθεση για τη στρατηγική καταπολέμηση της διαφθοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ καλό έγγραφο βάσης για να μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε καλύτερα το τοπίο της διαφθοράς σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να δούμε ποια είναι τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας για να αντιμετωπίσουμε καλύτερα το πρόβλημα αυτό. Χαιρετίζουμε την Επίτροπο κυρία Μάλστρομ και την ευχαριστούμε που είναι παρούσα εδώ σήμερα για να παρουσιάσει την έκθεση της Κομισιόν σε σχέση με τη διαφθορά και στη συνέχεια θα έχουμε συζήτηση. Καλώς ήλθατε κυρία Μάλστρομ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρίε και κύριοι. Αξιότιμα μέλη, χαρά μου που είναι εδώ ξανά. Και είμαι εδώ πρώτα απ' όλα για να παρουσιάσω την έκθεση να πάρει τη διαφθορά. Βέβαια, μπορώ να απαντήσω και σε άλλε ερωτήσει, εάν υπάρξουν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεχώ υποστήριζε το έργο κατά τη διαφθορά και την πρωτοβουλία. Θέλω να σα ευχαριστήσω πραγματικά για την υποστήριξή σα που παρήχατε και προ εμένα και προ το προσωπικό μου καθ' όλη τη διάρκεια τη θητεία. Συνεχώ όλε τι εκθέσει και στι συζητήσει αναφέρατε πώ η διαφθορά διαβρώνει την εμπιστοσύνη του κοινού στα, όσον αφορά τα δημοκρατικά θεσμικά όργανα, εμποδίζει την εσωτερική αγορά, τις επενδύσεις και ενθαρρύνεται το έγκλημα να βρει νόμιμους των εισαγωγικών τρόπους για να ξεπλύνει το χρήμα του. Ε, όλα αυτά αληθεύουν και βέβαια κοστίζει χρήμα των φορολογουμένων. Δισεκατομμύρια επί δισεκατομμυρίων το χρόνο. Το 2011 οι εκτιμήσεις, και είναι προσεκτική η εκτίμηση, είναι ότι το κόστος της διαφθοράς ήταν πάνω από 120 δις ευρώ το χρόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένας προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ενώσης. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε καιρούς λιτότητες αυτά τα χρήματα με άλλους τρόπους. Λοιπόν, είναι και, καινή η ώρα να εξεταστεί προσεκτικά η διαφθορά και με αυτή την έκθεση ε, κάνουμε αυτή την προσπάθεια επί μακρόν για να έχουμε την πιο καλή δυνατή έκθεση την ευθετή στην περασμένη εβδομάδα. Δίνει μια ειλικρινή αξιολόγηση στην κατάσταση σε κάθε 28 χώρε, πώ αντιμετωπίζουν τη διαφθορά, πώ οι φυστάμενοι νόμοι και οι πολιτικέ εφαρμόζονται, Αναφέρονται οι καλές πρακτικές, αλλά προτείνουμε και το πώς το κάθε κάτω μέλος μπορεί να βελτιώσει την προσπάθεια καταπολέμησης διαφθοράς. Η έκθεση δείχνει το επίπεδο της διαφθοράς, ποικίλει από χώρα σε χώρα μέλος, αλλά υπάρχει διαφθορά σε όλες τις χώρες. Δεν υπάρχει κάποια χώρα χωρίς διαφθορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οι πολίτες το ξέρουν και ανησυχούν. Δημοσιεύουμε επίσης ε, στοιχεία μέσω του Ευρωβαρομέτρου και δείχνει η βολιδοσκόπηση ότι πλέον 76% των Ευρωπαίων πιστεύουν ότι είναι ευρέω διαδεδομένη η διαφθορά στη χώρα του και πάνω από του μισού Ευρωπαίου πιστεύουν ότι το επίπεδο τη διαφθορά στη χώρα του έχει αυξηθεί. Είναι μια αντίληψη. Ε, ε, Αλλά είναι σοβαρή κατάσταση. Ένα από του 12 Ευρωπαίου ήταν ήδη μάρτυρα διαφθοράς την περασμένη χρονιά και περίπου 40% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που ζήτησαν πούμε, την άποψή του θεωρούσαν τη διαφθορά ότι αποτελεί εμπόδιο όσον αφορά το επιχειρήν στην Ευρώπη και βέβαια είναι σοβαρότατο αυτό. Υπήρξε σημαντική αύξηση όσον αφορά τις συζητήσεις απεσάστηκαν συζητήσει για την καταπολέμηση διαφθορά και οι πολιτικέ κατά τη διαφθορά συζητούνται εκτενώ σε πολλέ χώρε. Έχουν αποκτήσει προτεραιότητα και για τα κόμματα και για τα κινήματα. Ε, προέβαλαν τέτοια επιχειρήματα ε, και έχουμε νέες νομοθεσίες, νέους θεσμούς που δημιουργήθηκαν και διάφορες στρατηγικές καταπολέμησης διαφθοράς. Όλα αυτά είναι πολύ καλά. Ε, λαμβάνουμε υπόψη τις εξελίξεις και την πρόοδο και όπως σας είπα δείχνουμε ποιες είναι οι πολύ καλές πρακτικές που υπάρχουν σε διάφορες χώρες. Ταυτόχρονα όμως, όπως δείχνει και η έκθεση, αυτά δεν αρκούν. Τα αποτελέσματα δεν είναι αρκετά και αυτό λυθεύει για όλα τα κράτη-μέλη. Οι φυστάμενοι νόμοι και οι πολιτικές δεν εφαρμόζονται αρκετά καλά και δεν υπάρχει πραγματική πολιτική βούληση για την εκρίζωση της ε, διαφθοράς. Ανεπαρκής ε, κατανόηση των συνεπιών της διαφθοράς και έτσι δεν λαμβάνεται σε όλες τις πολιτικές υπόψη κατά τη διαφθοράς από τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων στην τοπική αυτοδιοίκηση, στι κρατικέ προμήθειε, δεν λαμβάνονται υπόψη. Θέλουμε να βελτιωθούν διάφοροι τομεί. Λοιπόν, θα μπορούσαν να είναι η χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε κάποια κράτη-μέλη που θα πρέπει να εξεταστεί. Σε άλλε χώρε το, ευάλ, το ε, ε, τον ευάλωτο χαρακτήρα που έχει διαφθορά όσον αφορά τι δημόσιε προμήθειε. Είναι ευάλωτο δημόσιε προμήθειε λόγω διαφθορά και οι δημόσιες ε, και η πρόσβαση στην υγεία επίσης. Πολλοί πρέπει να δίνουν φακελάκι για να έχουν περίθαλψη. Ε, βλέπουν ότι οι περισσότερες συστάσεις ε, αφορούν και τα 28 κεφάλαια, για κάθε χώρα δηλαδή. Συνετάχθη έκθεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την συμβολή πανεπιστημιακών, εθνικών εμπειρογνωμόνων, διεθνών οργανισμών κλπ. κλπ. Έγιναν διάφορα σεμινάρια και συζητήσεις με τους επαΐοντες συμπεριλαμβάνεται στην έκθεση μια επισκόπηση των διαφόρων τάσεων όσον αφορά τη διαφθορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβάνεται και θεματική προσέγγιση όσον αφορά τις δημόσιες και μετά έχουμε συγκεκριμένες αναφορές, συγκεκριμένα κεφάλαια για κάθε μία από 28 χώρες. Οι προτάσεις ποικίλουν από χώρα σε χώρα, αλλά υπάρχουν παραδείγματα όπως η ενίσχυση της δυνατότητας ε, ελέγχου των διαφόρων φορέων, ένα μεγαλύτερος έλεγχος διαφάνεια, η χρηματοδότηση των ε, πολιτικών κομμάτων, ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου, των δημοσίων αρχών, ενίσχυση συστημάτων αποκαλύψεως των πηγών ε, περιουσιακών στοιχείων, βελτίωση τη αποτελεσματικότητα των πολιτικών καταπολέμηση σύγκρουση συμφερόντων, εφαρμογή αποτελεσματικότερων πολιτικών για την καταπολέμηση τη διαφθορά σε τοπικό επίπεδο, κυρίω σε τομεί που είναι ευάλωτοι στη διαφθορά. Θέλουμε καλύτερη αποτελεσματικότητα των συγκελικών αρχών, των δικαστηρίων, των διοκτικών αρχών. Θέλουμε οι φορεί καταπολέμηση διαφθορά να είναι πιο ανεξάρτητοι, όπου υπάρχουν αυτοί, να εξασφαλίσουμε ότι διάφορε ποινικέ διώξει όσον αφορά τι ε, τη διαφθορά εκλεγμένων πολιτικών να μην καταπολεμούνται, να μην ποδίζονται να είναι αποτελεσματική ε, προστασία εκείνου που δίνουν πληροφορίε. Θα πρέπει να καταγράφεται που υπάρχουν δωροδοκίε, κυρίω στον τομέα τη άμυνα. Και πρέπει, χρειάζεται καλύτερα μέσα του ώστε να εξασφαλίζεται η διαφάνεια φορών ομάδε πίεση. Πρέπει να υπάρχουν μηχανισμοί και πολιτικέ για τη μετώπιση τη διαφθορά που σχετίζεται με εταιρείε που ανήκουν στο κράτο ή ελέγχονται το κράτο και χρειάζονται περισσότερα ηλεκτρονικά εργαλεία για μεγαλύτερη διαφάνεια και έλεγχο των δαπανών σε κυβερνητικό επίπεδο και σε τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτέ είναι κάποιε από τι συστάσει που περιέχονται στο κείμενο. Όπω προανέφερα, κοιτάξαμε εκ του συνέγγυε στις ε, δημόσιε προμήθειες, όπω γνωρίζετε, το 1 πέμπτον του ΑΕΠ τη Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε χρόνο ξοδεύεται τι δημόσιε αρχέ, κρατικέ αρχέ, όσον αφορά την προμήθεια αγαθών, υπηρεσιών και έργων ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τεράστια ποσά και 20% από αυτά αφορούν τι δημόσιε προμήθειε που ξεπερνούν ε, τα όριο που καθορίζεται για να εφαρμόζονται η κανόνε Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, Έκανε έρευνα η Όλαφ κατ' ομετήματο του Κοινοβουλίου και η έκθεση υπευρύθη πέσει τον Οκτώβριο και Όλαφ εκτίμησε το 2010 η διαφθορά όσον αφορά τι δημόσιε προμήθειε σε μόνο πέντε τομεί σε 8 κράτη-μέλη κόστησε ανάμεσα στο 1,4 και 2,2 δις ευρώ το χρόνο. Και σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, και την έκθεση του Ευρωβαρομέτρου τη περσμένη εβδομάδα, ένα τρίτο των εταιριών που συμμετείχαν σε δημόσιου διαγωνισμού είπαν ότι τι εμπόδισε ε, η διαφθορά από ανάθεση έργου ή να πάρουν σύμβαση. Οπότε πρέπει να γίνουν μεγάλε προσπάθειε στο κράτη-μέλη για να αποφευχθεί η διαφθορά στον τομέα των δημοσίων προμηθειών. Χρειάζεται συστηματική χρήση, πιο συστηματική χρήση τη αξιολογήσεω κινδύνου διαφθορά σε κάθε τομέα. Χρειάζεται εφαρμογή προτύπων υψή τη διαφάνεια όσον αφορά τον τομέα των διαγωνισμών και των προμηθειών καθώς και την ανάθεση έργων και υπογραφή συμβάσεων. Χρειάζονται μηχανισμοί εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου, καλύτεροι μηχανισμοί να γίνεται γενική επισκόπηση, μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση όσον αφορά την πρόληψη και χρειάζεται να επιβάλλονται αυστηρότερε κυρώσει όσον αφορά την παραβίαση κανόνων περί προμηθειών. Τι λεπτομέρειε τι έχετε στην έκθεση. Όλα αυτά είναι μια πρώτη αναφορά, είναι μια πρώτη έκθεση, μεγάλο βήμα που για πρώτη φορά έχουμε τέτοια έκθεση. Βέβαια είναι μόνο ένα πρώτο βήμα. Είναι σημαντικό διότι έχουμε σφαιρική εικόνα της καταστάσεως στα κράτη-μέλη και έχουμε και προτάσεις για περαιτέρω πρόοδο. Τώρα θα ακούσουμε τα κράτη-μέλη, εσάς βεβαίως, τα Εθνικά Κοινοβούλια, την Κοινωνία των Πολιτών και άλλους ενδιαφερομένους και θα συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη τους ώστε να δούμε πώς οι προτάσεις αυτές θα εφαρμοστούν. Και θα κινητοποιήσουμε φέτος ένα πρόγραμμα ανταλλαγή εμπειριών για να στηρίξουμε τα κράτη-μέλη με συμμετοχή διαφόρων εμπλεκομένων φορέων, και μη κυβερνητικών οργανώσεων για να εφαρμόσουμε τι προτάσει. Θα εξακολουθούμε τα θέματα καταπολέμηση διαφθορά, συμπεριλαμβάνουμε στη συνοχή, στι δημόσιε προμήθειε, στη διεύρυνση, αναπτυξιακή βοήθεια κλπ. και σε άλλε πτυχέ πολιτική να συμπεριλαμβάνουμε την καταπολέμηση διαφθορά. Και έχουμε δεσμευτεί να το κάνουμε νωρίτερα, ότι θα το κάνουμε, αλλά επιβεβαιώνει η έκθεση ότι υπάρχει η ανάγκη για πραγματικά μια ολιστική προσέγγιση τα επόμενα χρόνια. Επίσης θα ασχοληθούμε με την καταπολέμηση διαφθοράς κατά το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, οπότε χρειάζεται αυτό για να στηρίξουμε την οικονομική ανάκαμψη και χρησιμοποιήσουμε τα απορίσματα τη εκθέσεω για να αξιολογήσουμε τι περαιτέρω ανάγκε που υπάρχουν πρόθεσμα για θέσπιση νέα νομοθεσία, αν κάτι τέτοιο παραστεί αναγκαίο. Και βάσει όλων αυτών, σε δύο χρόνια θα υπάρξει επόμενη έκθεση που θα αναφέρεται σε όλα όσα θα έχουν γίνει και ελπίζουμε από την επιτευχθήσα πρόοδο που θα την πετύχουμε όλοι μαζί. Βέβαια, μια έκθεση δεν είναι ο μόνος τρόπος πολεμής διαφθοράς, αλλά είναι ένα εργαλείο και δεν μπορούμε να κολλησιεργούμε. Και προσβλέπω σε συζήτηση του θέματος αυτού μαζί σας και να προχωρήσουμε όσον αφορά τη συζήτηση και τη συζήτηση στα διάφορα κρατημέλη. Κύριε Πρόεδρε, να πω κάποια λόγια για ένα θέμα το οποίο συζητήσαμε επανειλημμένα και που οδήγησε σε πολλές γραπτές ερωτήσεις και επιστολές όσον αφορά το PNR, τα στοιχεία επιβατών. Ε, θα ήθελα να ξεκινήσω με την οδηγία για το PNR, την Ευρωπαϊκή όσον αφορά τα στοιχεία επιβατών. Ξέρετε ότι αυτό το θέμα αναπέμφθηκε στην Επιτροπή πέρσι τον ε, Ιούνιο και διεξήχθησαν συζητήσει στο άτυπο Συμβούλιο Εσωτερικών και Δικαιοσύνη πριν από δύο εβδομάδε στην Αθήνα, ήταν παρόν και ο Πρόεδρος και υπήρξε σχεδόν ομόφωνη έκκληση από πλευρά κρατών μελών από του υπουργού να σημειωθεί πρόοδο όσον αφορά την οδηγία και υποστηρίζουμε αυτή την έκκληση από πλευρά Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή. Εν τω μεταξύ, Αυξανόμενο αριθμό κρατών μελών δραστηριοποιείται σε εθνικό επίπεδο για να δημιουργήσει το δικό του σύστημα PNR με βάση εθνικό δίκαιο και αυτό επίση έχει σαν κίνητο τη σοβαρή απειλή που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, παραδείγματο χάρη από διάφορου Ευρωπαίου που πάνε στη Συρία να πολεμήσουν ε, οι αλλοδαποί πολεμιστέ και μπορεί έτσι μέσω PNR να δούμε ποιοι είναι οι ξένοι πολεμιστέ που φεύγουν την Ευρωπαϊκή Ένωση ή μέσω αεροπορικών συγκοινωνιών επιστρέφουν στην Ευρώπη οπότε οι δυνάμεις της τάξης ξέρουν ποια είναι η μεσω αεροπορικων συγκοινωνιων επιστρεφουν στην ευρωπη οποτε οι δυναμεις τη ταξης ξερουν ποια ειναι η προθεση των διαφόρων ατόμων να ταξιδέψουν και ετοιμάζονται καταλήλω. Λοιπόν, ε, δεν έχουμε PNR σε ευρωπαϊκό επίπεδο όμω. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμω παρέχει συγχρηματοδότηση σε κάποιε εθνικέ δραστηριότητε και το έχουμε καθορίσει αυτό και σε επιστολή προ τον Πρόεδρο, ούτω ώστε να προσπαθήσουμε να πετύχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή συνοχή μεταξύ εθνικών συστήματων και σε και θέμα υψηλότερο επίπεδο προστασία των δεδομένων. Έχουμε περιορισμένα μέσα όμω, χωρί να υπάρχει ε, ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία. Μόνο μια οδηγία ευρωπαϊκή για το PNR θα εξασφαλίζει ότι, ότι προστατεύουμε παρκώς τα στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρουμε ότι είναι πολύ ευαίσθητο θέμα αυτό, το θέμα των στοιχείων και η επεξεργασία των στοιχείων και στην Επιτροπή τη δική σα και στο Κοινοβούλιο. Ελπίζουμε να βρούμε μια διέξοδο για να καταπολεμήσουμε το σοβαρό έγκλημα και τρομοκρατία, όμω έχοντα ύψιστα επίπεδα ε, προστασία ε, των δεδομένων και ακαιρεότητα αυτή τη διαδικασία. Υπάρχει και θέμα PNR που σχετίζεται με τη Ρωσία και να σα πω ότι ήμουν στη Μόσχα πριν από 15 μέρε και η Ρωσική Ομοσπονδία μέσω του Υπουργού της επιβεβαίωσε απευθυνόμενο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ζητήσει στοιχεία PNR χωρίς ζητή συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αυτό θα κάνει η Ρωσική Ομοσπονδία θα είναι να χρησιμοποιήσει νομοθεσία API και θα ξεκινήσει αυτό τον Ιούλιο του 2014. Δυστυχώς θα συμπεριλαμβάνεται στον έλεγχο αυτό, θα συμπεριλαμβάνονται και υπερπτήσεις το PNR συζητείται και με το Μεξικό. Το Μεξικό θέσπισε νομοθεσία δική του για τη συλλογή στοιχείων επιβατών, την αναβολή της εφαρμογής της νομοθεσίας, μέχρι ότου να έχουμε διευθετήσει το ζήτημα από πλευρά Ευρωπαϊκής Ενώσεω. Είμαστε επαφή με τους Μεξικανούς ε, εταίρους μας. Συνάντησα τον Υπουργό των Αρμόδιων την περασμένη εβδομάδα. με την προσωπία στο Μεξικό τέλος ε, Μαρτίου, τόσο ώστε να το συζητήσουμε αυτό Ενθαρρύνουμε βεβαίως το Μεξικό επίσης να χρησιμοποιεί τα στοιχεία API και όχι σε πλήρες σύστημα PNR. Και τέλος, όσον αφορά το θέμα το θέμα του προγραμματισμού στα πλαίσια του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου έλαβα επιστολή από τον Πρόεδρο ζήτησα τον Γενικό Διευθυντή, τον κύριο Μοσχοβίτση, να παρουσιάσει μια επισκόπηση τη προόδου που έχει επιτευχθεί, να ενημερώσει την Επιτροπή σα. Όπω θα ξέρετε, επιμείναμε με την υποστήριξή σα αυτό το εγχείρημα είναι το διαφανέστερο δυνατό. Ο κ. Μοσκοβίτσι διεξήγαγε διάλογο με όλα τα κράτη-μέλη και θα δώσει όλες τις πληροφορίες σε εσά ούτως ώστε να είστε πλήρως ενήμεροι. Βέβαια διεξάγονται συζητήσεις σε υψηλό επίπεδο όχι πολιτικό. Θα σας ενημερώσει πλήρως λοιπόν σε μια καθορισμένη ημερομηνία. Θα συναντηθούμε με τη γραμματεία. Με όλα αυτά, ελπίζω, Πρόεδρε, να πάτε σε κάποιε ερωτήσει, αλλά βεβαίω είμαστε στη διάθεσή σα, ούτω ώστε να ακούσω σχόλια και ερωτήσει από τα αξιότιμα μέλη. Ευχαριστώ την προσοχή σα. Ευχαριστώ πολύ, Επιτροπή Μάλστρομ. Είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μα εκθέσατε. Κανείς δεν θα μπορούσε να τονίσει πόσο σημαντικό είναι το ζήτημα αυτό και για τα μέλη της Επιτροπής Θεμελιωδών Ελευθεριών αλλά και για τους Ευρωπαίους πολίτες. Γιατί πρέπει να εξασφαλίσουμε, να διασφαλίσουμε μάλλον ότι τα χρήματα των φορολογωμένων φτάνουν και χρησιμοποιούνται για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται και ότι η διαχείρισή τους είναι χρηστή. Η σημασία αυτή είναι ακόμα πιο σημαντική όταν μαθαίνουμε πόσο υπερβολικά, πόσο τεράστια είναι τα κόστη που προκαλεί η διαφθορά. Είναι επίσης σημαντικό να καταπολεμηθεί η διαφθορά, προκειμένου να υπάρχει εμπιστοσύνη των πολιτών και να μην θεωρούν ότι συμφέροντα που κρύβονται πίσω από κλειστές πόρτες στην πραγματικότητα μας επηρεάζουν στον τρόπο με τον οποίο αξιοποιούμε τα εξαιρετικά περιορισμένα χρήματα που έχουμε. Τώρα που έχουμε φτάσει να μετράμε και το τελευταίο σεντ. Κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης που έχει ήδη συμπληρώσει τέσσερα χρόνια. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στα μέλη του Κοινοβουλίου. Προβλέπεται λοιπόν συζήτηση μετά την παρουσίαση της Επιτρόπου. Έχω ήδη ε, σημειώσει ορισμένους. Η κυρία Άννα Ευχαριστώ την, ε, εκπρόσωπο, την Επίτροπο Μάλστρομ για αυτή την έκθεση την οποία αναμέναμε πέρυσι, αλλά είναι πολύ σημαντική, παραμένει πολύ σημαντική. Την διάβασα με μεγάλη προσοχή και ιδιαίτερα το κεφάλαιο που αναφέρεται στη χώρα μου, την Πορτογαλία. Και θα έλεγα ότι είναι ε, ορθός ο τρόπος και ακριβής ο τρόπος με τον οποίο εξηγεί το πρόβλημα. Αναφέρει ότι δεν υπάρχει στρατηγική, δεν υπάρχει ούτε μηχανισμός για την αντιμετώπιση της διαφοράς στην Πορτογαλία και επίσης αναφέρει ότι το 90% των πολιτών στην Πορτογαλία θεωρεί ότι η διαφθορά είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Κάτι το οποίο επιδεινώθηκε τα τελευταία τρία χρόνια. Τι έγινε τα τελευταία τρία χρόνια? Ήταν ακριβώς αυτά τα τρία χρόνια της υπαγωγής μας στην Τρόικα και το σχέδιο διάσωση. Ε, μια τρόικα η οποία παρεπιπτόντως να πούμε ότι συμπεριλαμβάνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το γεγονό λοιπόν ότι αυξήθηκε η διαφθορά αυτά τα τρία, τελευταία τρία χρόνια, μάλλον αυτή η αίσθηση, είναι μια αίσθηση την οποία τη μοιράζομαι και εγώ μαζί με όλου του υπόλοιπου πολίτες. Δεν είναι η Πορτογαλία που δεν έχει ε, ε, στρατηγική για την αντιμετώπιση της διαφθοράς, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά. Γιατί όπως λέει και η έκθεση η διαφορά δεν είναι κάτι που αφορά μόνο την Πορτογαλία ή ε, αφορά μόνο την Ελλάδα ή είναι ενδυμικό σε αυτές τις χώρες, είναι κάτι που αφορά και τη Γερμανία. Είναι ένα πρόβλημα που ε, έχει δημιουργηθεί στην Ευρώπη συνολικά επειδή έχουμε αφήσει ανεξέλεγκτο αυτό το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Έχει επιδονωθεί βεβαίως η κατάσταση στην Πορτογαλία τα τελευταία τρία χρόνια. Πώς θα τον αντιλαμβάνονται οι Πορτογάλοι πολίτε. Και αυτό εξαιτία ενεργειών που γίνονται υπό την αιγίδα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπω οι ιδιωτικοποιήσει στην Πορτογαλία, στην Ελλάδα και αλλού. Αυτέ οι ιδιωτικοποιήσει ήταν μία από τι σημαντικότερε πηγέ διαφθορά. Το μνημόνιο που συνοδεύει το ε, σχέδιο διάσωση δεν αναφέρει καν τη λέξη διαφθορά, δεν αναφέρεται καν η καταπολέμηση τη διαφθορά στο μνημόνιο δόθηκαν φορολογική δόθηκε φορολογική αμνηστία με τις ευλογίες της Τρόικας από την Πορτογαλική κυβέρνηση. Ε, αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για κάποιον ο οποίος έχει ε, ε, κέρδη ή χρήματα αποκτήσει με παράνομο τρόπο, είναι ο καλύτερος τρόπος με φορολογική αμνηστία για να τα νομιμοποιήσει. Του ζητάμε απλώς να πληρώσει ένα μικρό ε, ποσοστό 5% για να τα επαναπατρίσει χωρίς να ρωτήσουμε τίποτα σε σχέση με την προέλευσή του, Και αυτό έγινε με τις ευλογίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λοιπόν, εκτιμώ τι προσπάθειες που κάνετε και πράγματι θεωρώ την έκθεση σωστή και ε, διεξοδική. Πράγματι αναφέρει τα και τα προβλήματα και τι χρειάζεται να γίνει για να καταπολεμηθούν. Είπατε όμως ότι αυτά θα πρέπει να, να, να, να συμπεριλάβουμε στι αξιολογήσει που γίνονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Συμφωνώ βεβαίω, αλλά αυτά πρέπει να δημοσιοποιούνται επίση. Μίλησα για τη χώρα μου ω παράδειγμα μιας ε, κατάσταση και ενό προβλήματο που είναι πραγματικά ευρωπαϊκό. Στην ε, έκθεση σα αναφέρεστε σε κάποια συγκεκριμένες, συγκεκριμένα περιστατικά, συγκεκριμένες υποθέσεις στην Πορτογαλία. Σε μια υποσημείωση αναφέρετε τα υποβρύχια. Στην Ελλάδα, πάλι για παρόμοια υπόθεση, την υποβρύχια, από τα οποία πουλήθηκαν από γερμανικές εταιρείες, έχει ήδη ξεκινήσει μια έρευνα. Αλλά η Γερμανία δεν δίνει την δυνατότητα ανάκριση των ανθρώπων που δωροδόκησαν Πορτογάλους και Έλληνε αξιωματούχου στο πλαίσιο αυτών των υποθέσεων, γιατί έγινε μια συμφωνία. Και η εισαγγελία του μονάχου όταν απευθύνθηκα μου απάντησε αυτό. Έχει αποδειχθεί στην Πορτογαλία λοιπόν ότι υπήρξαν μίζες στο ζήτημα των υποβρυχίων και είναι κλασικό παράδειγμα δημοσίας προμήθειας στην οποία υπήρξε διαφθορά, η υπόθεση των υποβρυχίων. Τι έγινε λοιπόν σε αυτή την υπόθεση, οι πολίτες αισθάνονται ότι τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει, ότι οι πορτογαλικές αρχές συνέβαλαν καταλήγω στην, ε, στις συλλήψεις τελικά και στις φυλακίσεις στη Γερμανία, αλλά όσον αφορά τους Πορτογάλους δεν έγινε τίποτα. Κανείς δεν τιμωρήθηκε. Και γιατί αυτό, γιατί τυχαίνει ο υπεύθυνο, ο υπέτειος να είναι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Μπαρόζο. Και γι' αυτό κουκουλώθηκε το θέμα και η διαδικασία ε, καθυστερεί και κολλησιεργούμε. Κάθε φορά που ένα εισαγγελέα αντιλαμβάνεται τη δικογραφία και καταλαβαίνει τι έχει γίνει, τον αλλάζουμε για να μην μπορέσει να προχωρήσει την εξέταση και τη δίωξη τη υπόθεση. Ναι, εξαιρετική υπόθεση λοιπόν το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο για να εξετάζουμε τέτοιες υποθέσεις. Και να σας δώσω και μια άλλη υπόθεση που και πάλι αφορά τη Γερμανία, την Ελλάδα και την Πορτογαλία, πιθανώς και άλλες χώρες. Και είναι μια υπόθεση στην οποία η Επιτροπή φέρει ιδιαίτερη ευθύνη. Στην υπόθεση αυτή, η σημερινή Γουινέα, μία από τις πλέον διεφθαρμένες ε, κυβερνήσεις στον κόσμο, συν αποφάσισε να εξαγοράσει το κεφάλαιο μιας πορτογαλικής ε, τράπεζας που χρειαζόταν να διασωθεί. Τελικά όμως αυτά τα κεφάλαια πληρώνονται ε, μέσω του προγράμματος διάσωσης από τους Πορτογάλους φορολογούμενους και ήλπιζα τουλάχιστον σε αυτή την υπόθεση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ασκήσει το ρόλο της, όπως και η ΕΚΤ θα έπρεπε, έτσι ώστε να σταματήσει αυτή την προφανή ε, ε, παράνομη, τέλος πάντων συνειφασμένη με διαφθορά συμφωνία και να μην της επιτρέψει να συναυθεί. Ευχαριστώ κυρία Γκόμες για την ε, ε ένθερμη αυτή καταγγελία σας. Τώρα ο κύριο Τεγιόγκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την κυρία Επίτροπο για την παρουσία της εδώ. Νομίζω ότι το 2011 όταν είχαμε για πρώτη φορά άτυπες συζητήσεις και συνεδριάσεις για μια σειρά θεμάτων μαζί με άλλους ομοφρονούντες ε, ευρωβουλευτές είχαμε συλλέξει και είχαμε τα στοιχεία και ήμουν πεπισμένο από την αρχή ότι είχατε μια προσήλωση προς την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος και αυτό διαφαίνεται και από την έκθεση της Κομισιόν όπως ανέφερε και η κυρία Γκόμες είναι μια έκθεση που έχει πολύ ενδιαφέρον υλικό και μπορεί να διασταυρωθεί και με άλλες πηγές Εγώ δεν μπορούσα να βρω πάρα πολλά προβλήματα σε αυτά που λέει η Κομισιόν. Είναι λοιπόν έγκυρο αυτό το υλικό και χαιρόμαστε που μπορούμε να κάνουμε και αυτή τη συζήτηση. Εγώ τώρα κάνω ορισμένε παρατηρήσει να κάνω. Πρώτα απ' όλα, είδα κάπου στην έκθεσή σας ότι λέτε ότι η μικρή κλίμακα διαφθορά δεν είναι πια πρόβλημα και επίσης λέτε και έχετε δίκιο μάλλον ότι η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη εξακολουθεί να είναι πρόβλημα σε πολλές χώρες. Και ακόμα και πολλοί Ολλανδοί πολίτες έχουν πει ότι χρειάζεται για να πάρουν τις δημόσιες ε, υγειονομικές υπηρεσίες πρέπει να δώσουν και κανένα φακελάκι καμιά φορά και αυτό φυσικά δεν είναι απόλυτα αποδεκτό. Όλα αυτά λοιπόν που λέτε είναι πολύ σωστά, γιατί νομίζω πρέπει να εστιάσουμε όχι μόνο σε τέτοια θέματα, αλλά και σε θέματα δημοσίων προμηθειών. Για πολλούς πολίτες όμως, η διαφορά μικρής κλίμακος είναι ιδιαίτερα ορατή. Θα ήθελα λοιπόν να γίνεται πάντα αυτή η διάκριση μεταξύ από τη μία πλευρά της ε, μορφής αυτής διαφθοράς που είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη για τις δημόσιες προμήθειες, αλλά επίσης να έχετε και κάποια μνήμα για τη διαφθορά χαμηλού επίπεδου. Δεύτερον, και σωστά πιστεύω, η Κομισιόν ζητά από τα κρατημέλη να εφαρμόσουν πλήρω την οδηγία για την <clears throat> διαφθορά στον ιδιωτικό χώρο. Αλλά δεν νομίζω ότι μας έχετε δώσει πολλά στοιχεία σε αυτά στην ε, έκθεσή σας. Έχετε πάρα πολύ υλικό βέβαια η έκθεσή σας, πολλά παρατήματα, αλλά δεν λέτε πολλά για διαφθορά σε ιδιωτικό επίπεδο, δηλαδή δοσοληψίες ε, διαφθοράς μεταξύ επιχειρήσεων στον ιδιωτικό τομέα. Και εδώ δεν έχουμε τα κατάλληλα εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να καταδεικνύεται αυτή τη μορφή διαφθοράς όταν λαμβάνει η χώρα όταν υπάρχει συνεννόηση μεταξύ εταιριών και κάνουν κάποιες συναλλαγές κάτω από το τραπέζι με τρόπο ο δεν είναι νόμιμος. Για, ευρύτερα θέματα. Τα πρώτα δύο στοιχεία στον κατάλογο δράσης μας για το 2011 αφορούσαν τα ίδια τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν θέλετε να πείτε στα κράτη-μέλη τι να κάνουν για να αντιμετωπίσουν τη διαφθορά, θα πρέπει να έχετε καθαρίσει την δική σας αυλή πρώτα. Και σε αυτή την περίπτωση είχαμε μια περίπτωση με 7 ευρωβουλευτές, οι οποίοι κατα... κατηγορήθηκαν για το γεγονός ότι είχαν μια ε, σύγκρουση συμφερόντων. Υπήρχαμε μια τέτοια περίπτωση στο και επίση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ελεκτικό Συνέδριο έχει ερευνήσει το θέμα των ομάδων εμπειρογνωμόνων. Έχουμε λοιπόν ένα τεράστιο θεματολόγιο που πρέπει να αντιμετωπίσουν τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και εγώ θα ήθελα να σα παρακαλέσω να υπάρξει μια χωριστή έκθεση κάποια στιγμή για τα όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και για τι σχέσει του με τα κράτη-μέλη. Αυτό θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο και νομίζω θα το εκτιμούσε και η κοινή γνώμη. Ένα άλλο θέμα για τι οικονομικέ επιπτώσει και ακολουθώ την ίδια κατεύθυνση που ανέφερε και η Αναγκόμε για την ε, διαφθορά σε ορισμένε από τις χώρες του ευρώ. Αναφέρεται ότι στην Ελλάδα η κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί. Ότι η ειδική μονάδα κατά της διαφθοράς στην Ελλάδα ήταν βέβαια ενεργή με πρωτοβουλία της Τρόικας, αλλά εγώ είχα προβλέψει ήδη εκ των προτέρων ότι με μια τέτοια περιορισμένη προσπάθεια δεν μπορεί να αλλάξει κανείς τα πράγματα. Αλλά πώς βλέπετε εσείς τη δυνατότητα για τις χώρες αυτές να μπορούν να βγουν από αυτή την κατάσταση όπου η κρή οικονομία είναι το 1 τέταρτο, ή στην Ιταλία το 1 πέμπτο της οικονομίας και να μπορέσουν να γίνουν με την άποψη αυτή πλήρη μέλη της Ευρωζώνης. Για μένα αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό εγχείρημα και για το μέλλον τελικά. Νομίζω ότι είναι κάπως δύσκολο όταν πάρουμε τώρα την έκθεση, αλλά επίκυνται οι ευρωεκλογέ και αναρωτιέμαι τι μπορούμε να κάνουμε. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να προκύψει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα ψήφισμα για το θέμα αυτό, αλλά ξέρω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μεγάλο αγώνα και συνοστισμό να μπουν θέματα στην ημερήσια διάταξη του Μαρτίου. Δεν ξέρω λοιπόν αν έχετε εσεί κάποια πρόταση για το πώ θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε κι εμεί και την Κομισιόν να είναι σε προεξάρχουσα θέση στην ημερήσια διάταξη το θέμα αυτό και στο επόμενο επερχόμενο κοινοβούλιο οι ομοφρονούντες με μένα βουλευτές είναι πάντα έτοιμοι να το προωθήσουν αυτό το θέμα, όπως αναφέραμε και στην επιστολή προς εσάς, αλλά θα θέλαμε να έχουμε κάτι απτό και συγκεκριμένο να αφήσουμε στους επιγόνους μας. Κέρκοφ. Έχουμε μια ψηφοφορία σε λίγο. Ζητώ συγγνώμη που έχασα την παρουσίαση. Να αναφερθώ λίγο για τα θέματα που είναι στα όρια της διαφθοράς. Είναι δύσκολες οι αποδείξεις νομικά. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί που υπάρχουν στα κράτη-μέλη με ενδιαφέρουν και τα θέματα της σύγκρουσης συμφερόντων. Μας κατηγορούν πολύ συχνά. Μα κατηγορούμεθα για του υπολογισμού μα, για τη χρήση των χρημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Πάντα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα είναι διεφθαρμένα και συμπεριφέρονται έτσι. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα δαπανούν όλα τα χρήματα. Και εγώ στην εκλογική μου περιφέρεια λέω ότι κάτι δεν ισχύει. Τα περισσότερα χρήματα ούτως ή άλλως που συζητούμε δαπανώνται στις χώρες μας. Και πολλά από τα ερωτηματικά όσον αφορά τη δαπάνη αυτών των χρημάτων ε, δημιουργούνται στις ε, χώρες μας. Το εξής θέλω να θέσω λοιπόν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να είναι πολύ πιο αυστηρή όσον αφορά τον εντοπισμό των προβλημάτων. Διαφορετικά πάντα ο κόσμος αυτή την άποψη θα έχει. Δηλαδή ανεξάρτητα από αυτά που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εξαλείψει τη διαφθορά, ανεξάρτητα από τι κάνει για να επιμένει επί των ελέγχων και να αντιμετωπίσει το θέμα συγκρούσεων συμφερόντων, πάντα θα ακούγεται αυτή η κατηγορία. Και είναι πολύ επικοδομητική η προσπάθεια σίγουρα και στη χώρα μου που θεωρείται ότι έχει πολύ ψηλά πρότυπα κατά τη διαφθορά. υπάρχουν πολλές ε, αδυναμίες όσον αφορά τα συστήματα εφαρμογής του νόμου. Έχουμε χάσει χρήματα και πόρους από την Ευρώπη επανειλημμένα. Υπάρχει πρόβλημα στον αφορά την ε, απορρόφηση των χρημάτων. Άρα αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσετε αν έχει την καλοσύνη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν μπορείτε να με καθησυχάσετε τελικά όσον αφορά αυτό. Ευχαριστώ η κυρία Γκυγιώμη έχει το λόγο. Ακόμα πιο γρήγορα, για να δώσω το χρόνο να απαντήσει η Επίτροπος, να πω κάποια λόγια. Αρκετά ενημερωτικά τα στοιχεία, όπως είπατε, αναφερθήκατε και ότι οφείλεται και στην αντίληψη που έχουν οι πολίτες. Το είπατε επανειλημμένα. Υπάρχει διαφορά μεταξύ αντίληψη και πραγματικότητας, ελπίζω τουλάχιστον. Ε, εν ώψη της μελλοντικής εκθέσεως. Τα κριτήρια προσμέτρησης, υπολογισμού, πώς θα δημιουργηθούν, θα έχουν επιστημονική βάση. Ούτω ώστε να υπάρχουν κριτήρια για τη συλλογή στοιχείων από το, που δημοσιεύονται στο ευρωβαρόμετρο άλλο ερώτημα για το κεφάλαιο για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα προβλέπετε να εξεταστούν επίσης και τα θέματα αυτά υποθέσεις διαφθοράς εντός των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπρόντς. Ευχαριστώ. Η παρουσίασή σας όμως πέρασε, μίλησε για θέματα πολύ ευρύτερα από την διαφθορά στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Μήπως θα έπρεπε καλύτερα να περιορίσουμε τον ορισμό της διαφοράς με τα θετικά κίνητρα που δίνονται για συγκεκριμένου τους επενδύσεις ή επίσης και για απειλές, για παράδειγμα την αποκάλυψη στοιχείων. Για παράδειγμα, το, το γεγονό ότι αποκαλύπτει ότι ένα πολιτικό έχει ένα συγκεκριμένο στυλ ε, ζωή που τον καθιστά ευάλωτο. Σε κάποιες χώρες χρησιμοποιούνται οικονομικά κίνητρα, δηλαδή δωροδοκίες ουσιαστικά, για να ε, επηρεαστεί η άποψη επιλογή κάποιου ατόμου ή μιας ε, κυβέρνησης. Είναι κάτι το οποίο έχει συμβεί στο Ηνωμένο Βασίλειο εδώ και ε, μάλλον 10 χρόνια πριν. Δεν πρόκειται να κάνω περιπτωσιολογία, δεν έχει νόημα σε ένα συγκεκριμένο περιστατικό πριν 10 χρόνια ένας δωρητής είχε κάποιες επαφές με μια χώρα με την οποία, η οποία είχε μάλλον κάπως ε, αμφισβητούμενες ε, σχέσεις με τους, γειτον, με τους γειτονές της και είχε χρηματοδοτήσει όλα τα πολιτικά κόμματα για να προωθήσει τις θέσεις του. Εγώ προσωπικά θεωρούσα ότι πάντοτε αυτό ήταν ε, μια προσπάθεια διαφθοράς. Εδώ δεν προσπάθησε αυτός ο άνθρωπος να κερδίσει κάτι, απλώς προσπάθησε να εξαγοράσει την υποστήριξη πολιτικών κομμάτων. Κάτι ακόμα. Η διαφθόρα μερικές φορές είναι τόσο υπόγεια που μερικές φορές είναι δύσκολο να την καταδείξει κανείς. Για παράδειγμα προσκλήσεις ή ε, κοινωνικές εκδηλώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επηρεάσουν κάποιον που λαμβάνει υποφάσεις. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που λαμβάνουν αποφάσεις θα μπορούσαν να εκπαιδευτούν για να μην ε, δέχονται πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να δημιουργήσουν την λαθασμένη εντύπωση ότι επηρεάζονται. Εγώ προσωπικά ποτέ δεν είχα υπάρξει ε, αντικείμενο τέτοια προσέγγισης. Ευχαριστούμε πολύ. Θα είμαι και εγώ πολύ σύντομη. Έχω μία ερώτηση. Αφού πρώτα ευχαριστήσω την Επιτρόπο Μάλστρομ για την ε, έκθεσή της και για το γεγονό ότι παρευρέθη για να μας την παρουσιάσει. Πράγματι, εργαστήκατε σκληρά για να προετοιμάσετε αυτή την εκθέση. Την διάβασα προσεκτικά, κρατώντας σημειώσεις. Υπάρχουν κάποια κράτη, ε, ε, ε, μέλη, η Βουλγαρία και η Ρουμανία, αρκετά χρόνια μετά την ένταξή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελούν στόχο ενός μηχανισμού ελέγχου της ε, διαφθοράς τους. Ενώ από την έκθεση προκύπτει ξεκάθαρα ότι η Βουλγαρία και η Ρουμανία δεν ε, είναι χώρες στις οποίες υπάρχει ιδιαίτερα μεγάλη διαφθορά ή ιδιαίτερα περισσότερο από τις υπόλοιπες χώρες. Επομένως, ποιος είναι ο λόγος που συνεχίζουμε να βρισκόμαστε στο στόχαστρο και τι μέτρα σκοπεύει να λάβει η Επιτροπή για να αντιμετωπίσει το ζήτημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο συνολικά. Ευχαριστώ. Ο κύριος, ο Μούλτερ ήταν στον κατάλογο επίσης. Έχετε το λόγο. Συγγνώμη, εγώ δεν μπορώ να σχολιάσω τα αρχικά λόγια της κυρίας Επιτρόπου γιατί δεν είμαι παρόν, αλλά παρακολουθώ τα νέα στις εφημερίδες και πρέπει να πω ότι είναι μια αξίεπαινη προσπάθεια της Κομισιόν. Θα πρέπει κάθε χρόνο να γίνεται αυτή η έκθεση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό εγχείρημα. Ένα θέμα το οποίο αναφέρθηκε προηγουμένως είναι το θέμα των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Νομίζω ότι αυτό είναι μια παράληψη ή αλλιώς την εντύπωση ότι είναι πεντακάθαρα τα ευρωπαϊκά όργανα, κάτι το οποίο είναι αμφισβητήσιμο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ελέγχει την Κομισιόν, οπότε αν η Κομισιόν ελέγχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ίσως υπάρχει μια δύσκολη σχέση. Πιστεύω όμως ότι στο μέλλον θα είναι καλύτερα για το ευρύ κοινό, για την κοινή γνώμη, αν αντιμετωπίζουμε όλο τον κόσμο και τα ευρωπαϊκά όργανα μαζί με τον ίδιο τρόπο. Λοιπόν, τώρα θα πάρουμε την απάντησή μας από την Επίτροπο Μάλστρομ. Να σας υπενθυμίσω ότι πράγματι αυτή η έκθεση είχε αντίκτυπο σημαντικό σε πολλά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ευλόγως. Υπάρχουν πολλές φορές ε, ορισμένες ε, ιδέες ε, οι οποίες κυκλοφορούν, οι οποίες είναι μια μορφή κοινοτυπιών και οι οποίε δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Πιστεύουν δηλαδή περικοί ότι η διαφθορά βρίσκεται μονάχα σε μερικέ χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, στι νέε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Όχι, η διαφθορά βρίσκεται παντού. Η κίνδυνη τώρα του να μην αντιμετωπίσουμε την διαφθορά αποτελεσματικά είναι πολύ μεγάλη και πρέπει να του λάβουμε στα σοβαρά. Δεν πρόκειται λοιπόν για την Α ή τη Β χώρα. Είναι για όλου μα ένα θέμα και ο κόσμος θεωρεί ότι η διαφθορά αυξάνεται και αυτό είναι εύλογο πάλι γιατί οι πολίτες ενοχλούνται όλο και περισσότερο για την αύξηση των ανισοτήτων που βλέπουν και τις θυσίες που τους επιβλήθηκαν. Από τον τρόπο με τον οποίο έγινε η διαχείριση της κρίσης και επίσης υπάρχει μια έρευνα που αφορά την συγκριτική ανάλυση εργαλείων και μέσων που είναι στη διάθεσή μας αλλά δεν νομίζω ότι είναι στο ύψος των προκλήσεων που έχουμε ενώπιον μας. Θα πρέπει, πιστεύω, να καινοτομήσουμε και να τολμήσουμε να, κάνουμε, να δημιουργήσουμε νέα εργαλεία που βρίσκονται στο ύψος των αρχών μας. Κάποια από αυτά είναι στο επίπεδο του εφικτού, όπως είναι το θέμα του εισαγγελέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και οι κοινέ προσπάθειες για το ποινικό δίκαιο και την εναρμόνισή του σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι σημαντικά. Όλα αυτά πρέπει να τα αναμένουμε για την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το επόμενο μάλλον, το οποίο θα πρέπει <clears throat> να είναι ακόμα πιο κοντά στις ανησυχίες του Ευρωπαίου πολίτη αν θέλει πράγματι να δώσει μια απάντηση στις ανησυχίες του, του Ευρωπαίου πολίτη και αυτή θα πρέπει να είναι η πρώτη απάντηση που θα δώσουμε μετά τις εκλογές του Μαΐου. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους για τα σχόλια και τις ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ γιατί μας στηρίξατε ένθερμα στην όλη διαδικασία της συντάξης εκθέσεως. Έπρεπε να είχε υποβληθεί νωρίτερα, απεδείχθη δυσχερέστατο εγχείρημα να βρούμε τη σωστή ισορροπία, να μην τονίσουμε ξεχωριστές ε, υποθέσεις, να βρούμε τις κατάλληλες δομές και τα ευάλωτα σημεία κάθε χώρας. το εγχείρημα. Η ομάδα μου έκανε πολύ αξιοσημείωτη δουλειά. Ήταν χρονοβόρα όμως και μάθαμε πολλά στη διαδικασία. Ήδη είδαμε πολλές συνέπειες αυτού, όχι μόνο στα μέσα ενημέρωσης. Έλαβα εκατοντάδες επί εκατοντάδων επιστολών από διάφορους πολίτες που μου στέλνουν καταγγελίες για υποθέσεις διαφθοράς και θέλουν να συμμετάσχουν στην προσπάθεια. Πολλά κράτη-μέλη θα σε επαφή μαζί μας και θέλουν ε, διάλογο μαζί μας. Και βέβαια και αιρετοί εκπρόσωποι από τοπικά κοινοβούλια και εθνικά κοινοβούλια θέλουν να συμμετάσχουν και θα πρέπει να οικοδομήσουμε πάνω σε αυτή την επιθυμία και ο εντατικό διάλογο με όλου είναι σημαντικότατο. Να δούμε πώ μπορούμε να δώσουμε συνέχεια. Ανεπίσημα και επίσημα. Οι δημόσιε προμήθειε επελέχθη στο βασικό θέμα για φέτο, ίσω του χρόνου. Την επόμενη φορά θα είναι ιδιωτικό τομέα, μικροδιαφθορά, ο τομέα τη υγεία. Θέλαμε ένα θέμα να τονίσουμε, όπου υπήρχαν και πολλά στοιχεία. Και έτσι μπορούσαμε να προβάλλουμε σαφέστερα επιχειρήματα. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έχουν μείνει εκτός, έχετε απόλυτο δίκιο όλοι σας που λέτε ότι έπρεπε να συμπεριληφθούν. Αυτή ήταν η πρόθεσή μας. Αυτή ήταν η αρχική μου πρόθεση και είχαμε ετοιμάσει τη σύνταξη σχετικού κεφαλαίου. Ήταν όμως δυσκολότατο να αυτοαξιολογηθούμε σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αναπόφευκτα το κεφάλαιο θα ήταν πολύ αδύνατο. Δεν μπορούμε να αυτοαξιολογηθούμε, πρέπει να δούμε τι κάνει το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Πρέπει να βρούμε κοινό έδαφος για την προσέγγιση. Ένα ανεξάρτητος φορέα θα μπορούσε να το κάνει. Ίσως θα μπορούσαμε να βρούμε κάποια λύση. Ε, μπορούμε να το συζητήσουμε μαζί. Πώς μπορούμε με αξιόπιστο τρόπο να κινηθούμε, να γίνει από ανεξάρτητο φορέα, ούτω ώστε το έγγραφο να είναι πραγματικά σοβαρό. Πρέπει να είμαστε ταπεινοί. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα δεν είναι απαλλαγμένα από τη διαφθορά. Πρέπει να δούμε τι βελτιώσει μπορούμε να επιφέρουμε, ποιε πρακτικέ μπορούν να εφαρμοστούν. Πώ μπορείτε να το υποστηρίξετε αυτό. Ξέρω ότι τελειώνει ο χρόνο, τελειώνει η θητεία. Μπορείτε να σα αποφασίσετε στο ψήφισμά σας για τη διαδικασία της Στοκχόλμης, αν εκεί μπορείτε κάπως να ενθαρρύνετε τη μελλοντική Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να δώσουν συνέχεια στην προσπάθεια. Εξετάζουμε τους ελεγκτικούς μηχανισμούς που καμιά φορά υστερούν, τους λείπει κοινοτικό χρήμα, το αναφέρεται, το είπαν και διάφορα κράτη-μέλη αυτό. Προς την κυρία Κιγιόμ λέω ναι ότι κοιτάμε ποιες αντιλήψεις υπάρχουν. Βέβαια είναι υψηλότερη εντύπωση από το πραγματικό επίπεδο τη διαφθορά. Και καμιά φορά ο κόσμο απογοητεύεται από του πολιτικού και προβάλλει τη διαφθορά σε υψηλότερο επίπεδο. Όταν του ρωτάμε, εσεί ε, δολοδοκίσατε, σα ζητήθηκε να δολοδοκίσετε, το είδατε με τα μάτια σα, για να έχουμε πιο ακριβεί πληροφορίε του χρόνου θα έχουμε και στατιστικά στοιχεία για το έγκλημα, συγκρίσιμα στοιχεία για όλα τα κάτι μελη και η διαφθορά είναι ένα από τα θέματα. Οπότε θα έχουμε και τα στοιχεία για την επόμενη έκθεση, θα έχουμε πραγματικά στοιχεία για τη διαφθορά με βάση την δίωξη στα... και την εκδίκαση υποθέσεων. Ο ορισμός κατάχρηση εξουσίας για ιδιωτικό κέρδος, κύριε Μπρόντς, αυτός είναι ο ορισμός που χρησιμοποίησαμε για τη διαφθορά και είναι ο ορισμός του ΟΗΕ είναι ευρύ ορισμός, αλλά γενικώ αποδεκτός, χρησιμοποιείται από πολλούς πανεπιστημιακούς επίσης. Θέτουμε θέματα δωροδοκία, ε, ομάδων πίεσης, χρηματοδοτήσεως, ε, πολιτικών κομμάτων, υπάρχει έλλειψη διαφάνειας και είναι ένα πρόβλημα που ανακύπτει πανηλημμένα. Λοιπόν, ο μηχανισμός, ο άλλο ο CBM που αναφέρατε είναι κάτι παράλληλο, δεν μπορώ να το ελέγξω εγώ. Αλλά όσον αφορά τη διαφθορά, υπάρχουν θέματα σε πολλές χώρες, πρέπει να εξεταστούν. Πρέπει να κάνουμε συγκρίσεις, πρέπει να μάθουμε ένας από τον άλλον. Όπως σας είπα, είναι ένα πρώτο σημαντικό βήμα αυτό. Τις επόμενες εβδομάδες θα προσπαθήσουμε να καθορίσουμε πώς θα δώσουμε κάποια συνέχεια, διότι δεν παρετούμεθα, δεν κλείνει το θέμα, έχουμε ενόψει την δεύτερη έκθεση και θα πιέσουμε τα κράτη-μέλη πάνω σε αυτό. Θα συζητηθεί στο Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών σε περίπου 15 μέρες, θα παρουσιάσω το θέμα. Έχουμε έρθει σε επαφή με πολλά κράτη-μέλη και κάποια κοινοβούλια πώς θα δώσουμε συνέχεια στη στάση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που με επιτρέψατε να έρθω και να παρουσιάσω το θέμα. Ευχαριστώ για την υποστήριξή σας και προσβλέπω σε συνέχιση του διαλόγου με τα παρόντα μέλη και τα άλλα μέλη του Κοινοβουλίου. Σε ευχαριστώ Επίτροπο Μάλστρομ, πολύ χρήσιμα αυτά που μας είπατε. Ήταν πολύ καλό αυτό, καλή παρουσίαση της πρώτης εκθέσεως της διαφθοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζουμε ότι θα ακολουθηθεί έκθεση από άλλα βήματα που θα βελτιώσουν την τωρινή κατάσταση. Χρειάζεται η προσπάθεια όχι μόνο αναλυτική και ελεγκτική, και για το πώς αντιλαμβάνεται ο κόσμος τη διαφθορά που χρειάζεται γι' αυτό να έχουμε κοινέ προδιαγραφές και κλείνει το μικρόφωνο του Πρόεδρου Hopefully making a difference. και ελπίζουμε να κάνουμε τη διαφορά τα επόμενα χρόνια για να μειωθεί η όλη εικόνα της διαφθοράς να μειωθεί η διαφθορά λόγω αποτελεσματικής καταπολέμησης λόγω καταστολής της διαφθοράς Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε Μάλστρομ τελειώσαμε Βλέπω να καταφθάνουν μέλη για την ψηφοφορία. Λοιπόν, προχωράμε για την ψηφοφορία. There will be Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, έτσι ώστε όλα τα μέλη να καθίσουν και να ετοιμαστείτε με τις ηλεκτρονικές σας κάρτες. Πέντε λεπτά διάλειμμα λοιπόν και επιστρέφουμε. Σας ευχαριστώ συνάδελφοι. Είμαστε έτοιμοι. Για καθίστε όλοι παρακαλώ. Ετοιμαστείτε παρακαλώ, ετοιμάστε τις ηλεκτρονικές κάρτες ψηφοφορίες και καθίστε. Και όσοι βρίσκονται στην αίθουσα, σας ζητώ την προσοχή σας, καθίστε και παραμείνετε ήσυχοι παρακαλώ γιατί η ψηφοφορία που έχουμε μπροστά μας θα μας πάρει λίγη ώρα, δεν είναι απλή. Ψηφίζουμε λοιπόν το προσχέδιο έκθεσης του εισηγητή μας, του κ. Κλοντ Μωράης, για το πρόγραμμα παρακολούθησης τη Υπηρεσία Εθνική Ασφαλεία των Ηνωμένων Πολιτειών, ε, του οργανισμούς παρακολούθησης διαφόρων κρατών μελών και τον αντίκτυπό του στα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώ και στη διατλαντική συνεργασία στον τομέα τη δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων. αυτό είναι ο τίτλο τη έκθεση. Ξεκινούμε λοιπόν. Ω συνήθω θα ακολουθήσω την, το κατάλογο ψηφοφορία για τι τροπολογίε, Και όταν χρειάζεται θα κάνουμε και ηλεκτρονική ψηφοφορία. Συμβαστική 1 υπέρ.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 Πέρας ψηφοφορίας. Προσθέτουμε μία ψήφο στους σοσιαλιστές. Όχι, μάλλον υπάρχει ένας ε, ψήφος παραπάνω στους σοσιαλιστές. Όχι, όλα σωστά τώρα. Και πέρας τις τώρα πάτε. Πέρας 25 υπέρ, 22 κατά, εγκρίνεται. Και τρεις αποχές. Για να το δούμε τώρα. Ζητά ε, κύριος Μιχέλε, ε, Ζητώ συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, αλλά περιμένω την, ε, ψηφοφορία, συγγνώμη, την κάρτα μου για την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Επομένως, ο Πρόεδρος προσθέτουμε άλλη μία ψήφο στις υπέρ, αλλά δεν αλλάζει το αποτέλεσμα. Λοιπόν, ψηφίζουμε τώρα τη συμβιβαστική 6 υπέρ Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 151 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 152 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 153. Ας ελέγξουμε αφού μου το ζητάτε. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 152. Παρακαλώ ψηφίστε. Πέρασε ψηφορίας. Και πάλι υπάρχει μία ψήφος παραπάνω από τους σοσιαλιστές. Ωραία, διορθώθηκε. 20 υπέρ 33 κατά απορρίπτεται. Ψηφίζουμε για την 152 υπέρ ε, ε, ζητά συγγνώμη ο πρόεδρος. 153. 153, συγγνώμη. 153. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ζητάτε έλεγχο. Θέλετε να ελέγξουμε την 153, αλήθεια. Καλά. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τροπολογία 153. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρασε ψηφοφορίας.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 Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και πηγαίνουμε στην τροπολογία 178. 178 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 179 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 180 υπέρ. Κατά. αποχές. Μου φαίνεται ότι απορρίφθηκε, αλλά ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά για να είμαστε σίγουροι. 180. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την 180. Παρακαλώ ψηφίστε. Και πάλι μια ψήφος παραπάνω στους ελιστές. Διορθώθηκε. Πέρα ψηφοφορία. 15 υπέρ, 38 κατά απορρίπτεται. 181 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 182 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ζητάτε έλεγχο βεβαίως. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 182. Παρακαλώ ψηφίστε. Πέρας ψηφορίας. Ναι, απορρίπτεται. 185 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 183 υπέρ. Κατά. Δεν είναι ξεκάθαρο. Διανατάσσεω χειρό. Σα ζητώ να σηκώνετε ψηλά τα χέρια σα για να είμαστε σίγουροι. Ηλεκτρονικό έλεγχο για την 183. Παρακαλώ ψηφίστε. Γιατί δεν ήταν σαφές. Πέρας φορές. Φυσικά τώρα είναι σαφές, 34 κατά, 17 υπέρ. Σας παρακαλώ να σηκώνετε ψηλά τα χέρια σας για να είναι πιο ξεκάθαρα τα αποτελέσματα. Θα διευκολυνθούμε όλοι. Συμβιβαστική 14. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 15. Η γραμματεία επισημαίνει ένα πρόβλημα στον πρόεδρο. Υπάρχει το ένα μέρος, το πρώτο μέρος της τροπολογίας 188. Γι' αυτό πρέπει να τεθεί σε ψηφοφορία. Το πρώτο μέρος της τροπολογίας 188. Διόρθωση. Για το δεύτερο μέρος πρέπει να ψηφίσουμε, λέει ο πρόεδρος. Λοιπόν, δεύτερο μέρος της 188 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτωκε. Συμβαστική 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Σύμβαστική Συμβιβαστική 16. Τμηματική ψηφοφορία για το πρώτο τμήμα. Η πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εκρίνεται Δεύτερο τμήμα υπέρ. Αποχέ, Εγκρίνεται. Να τα ελέγξουμε, να ελέγξουμε. Για το δεύτερο τμήμα τη συμβιβαστική 16 ψηφίστε παρακαλώ. against. 34 υπέρ 23 κατά εγκρίνεται. Άρα. Πηγαίνουμε στην τροπολογία 197 και την 211, οι οποίες είναι ταυτόσιμες. Έχουν το ίδιο κείμενο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Επόμενο. Ε, συμβαστική 17 υπέρ. Τι ζητάτε, δεν σας ακούω λέει ο Πρόεδρος. Κυρία Ματσέο, τι θέλετε. Θέλετε ηλεκτρονικό έλεγχο για την τελευταία ψηφοφορία λοιπόν. Ωραία. Εκτός μικροφώνου, πρόεδρος. Θα επαναλάβουμε την προηγούμενη ψηφοφορία ηλεκτρονικά για την 197-211 παρακαλώ ψηφίστε. τη ψηφοφορίας. «35 υπέρ 22 κατά εγκρίνεται». Προχωράμε λοιπόν. Συμβαστική 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2-13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2.14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 2.15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται 2.16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται 2.17 υπέρ. Κατά. Αποχές ε, απορρίπτεται. 2.18 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2.19 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2.20 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2.21 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 17α υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμ... Συμβιβαστική 18. Συμβαστική 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα. 2.24 και 2.25 μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Συμβαστική 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Όχι. Τροπολογία 2.28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 21 λέει ο πρόεδρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ναι, γιατί είναι συμβαστική 21. Και πάλι η γραμματεία επισημαίνει ένα λάθος στον πρόεδρο. Ζητώ συγγνώμη πρόεδρο, έχουμε περάσει την τροπολογία 2.31 και 2.32. Ψηφίζουμε για την 2.31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2.32 υπέρ. κατά αποχές απορρίψετε. Και πάλι συμβαστική 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2.36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 22 υπέρ. Μήπως θέλετε να αλλάξουμε. Μου ζητάτε να ελέγξουμε. Ωραία. Ελέγχουμε την τροπολογία 237. 237 παρακαλώ ψηφίστε. Πέρασε ψηφορίες. 32 υπέρ, 25 κατά και μία αποχή εγκρίνεται. Πηγαίνουμε λοιπόν τώρα στην συμβιβαστική 22 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 240 υπέρ, Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2.41. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2.43. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 242. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 246 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 245 να ελέγξουμε λέτε. Ωραία, ελέγχουμε την τροπολογία 246 έναρξη ψηφορίας. Λήξη ψηφορίας. 24 υπέρ, 32 κατά, απορρίπτεται και πηγαίνουμε στην 245 τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2044 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 247 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 248 υπέρ. Ζητά συγγνώμη. Έχει αποσυρθεί 252 λέτε. Γιατί 248 δεν πρέπει να ψηφίσουμε, ρωτά ο Πρόεδρος. Α, κατάλαβα, είναι ταυτόσιμη. Άρα, καταπίπτουν διάφορες και φτάνουμε στη 251. 251, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2.49 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2.50 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2.55 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2.59 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.58 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.61 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.63 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική 23 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 269 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 270 υπέρ. Να ελέγξουμε τη 269. Πάμε. Ζητήσατε έλεγχο, έτσι δεν είναι. Ωραία. Ελέγχουμε τη 269. Άρχεται. Πέρασε. Πέρας. 33-25 εγκρίνεται. 2,70 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 2,71 υπέρ. Κατά. Δεν είναι σαφές. Πάλι έλεγχος γιατί τη 2,71. Άρχεται. Άρχεται. Πέρασε. 28-27. Τσίμα τσίμα. Αλλά περνάει. 2.72. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2.82. Υπέρ. κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2,79 υπέρ. 2,77 προηγουμένως λέει ο πρόεδρος. Την ξέχασα. Συγγνώμη. 2,77. Κατά. Δεν είναι σαφές. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 2,77 άρχεται. περας 25.32 25-32 απορρίπτεται σαφώ. 2,79 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2,80 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2,81 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 2.83 έχει αποσυρθεί, 2.84 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται, 2.85 υπέρ. Έλεγχος ζητείτε για τη 2.84. Άρχεται. Πέρας. 32.26 εγκρίνεται. 2.85 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.86 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.87 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστή 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστή 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 302 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται απορρίπτεται απορρίπτεται Τριακόσια υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστή 27 υπέρ κατά αποχές δεκτή, συμβαστή 28 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 315 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, συμβαστική 29 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 322 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 323 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 324 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 325 υπέρ έλεγχος για την 324 324 άρχεται η ψηφοφορία πέρας 2532 απερίφθη. 326 λέει ο πρόεδρος. Συγγνώμη. 325 πρώτα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 326 υπέρ. Κατά. Αποχές Σύμβαση και 30 υπέρ. κατά αποχές δεκτή. 3.30 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 3.31 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 3.32 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 3.33. Α, απορρίπτεται, απορρίπτεται. 3.33 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 3.34 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 3.36 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 3.30 απορρίπτεται είπα. Έλεγχος. Θέλετε. Ε, καλά, να κάνουμε έλεγχο. 3.36. Έλεγχος. Πέρας. 21-35 απορρίπτεται 3-3-5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 3-37 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 31 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 340 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 341 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 32 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 33 υπέρ Θέλετε έλεγχο στην 32, συμβαστική. Εντάξει. «32 συμβαστική με ηλεκτρονικό έλεγχο. Άρχεται. Συμβαστική 32. Συμβαστική 32 ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 32-25. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 354 υπέρ. Κατά. Αποχές. 3 355 υπέρ. Κατά. Αποχές απολύπτεται. Συμβαστική 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. τη και 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 367 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 369 368 προηγουμένως Σπαρταράει ακόμα η 368. 368. Υπέρ. Κατά. Αποχέ, εγκρίνεται. 369. Υπέρ. Κατά. Αποχέ, απορρίπτεται. 370. Υπέρ. Έλεγχο για 369. Άρχεται. Άρχεται. Άρχεται η ψηφοφορία για την 369. περας 3621 εγκρίνεται. Εγκρίνεται. 371. Εκπίπτει. Συμβιβαστική 36. υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. 371, όχι αυτή εκπίπτει τώρα. Συμβαστική 36 υπέρ. κατά αποχές σύμβασης και 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 379 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 380 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 381 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 38 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 39 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 40. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 403 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 421 υπέρ κατά δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα επαναλαμβάνω 421 υπέρ κατά αποχές Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά θα κάνουμε έλεγχο. 4.21 τώρα, ηλεκτρονικός έλεγχος. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Έλεγχος. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται, πράγματι. 422 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 423 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 424 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 42 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 383 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 429 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 430 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 431 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 432 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 442 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 449 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 450 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 451 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 452 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 453 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 454 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 48 συμβαστική 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 49 σε, κατά τμήματα πρώτο τμήμα συμβαστική 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 460 λάθος λέει πρώτα συγγνώμη 466 466 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 50 υπέρ συγγνώμη έχουμε κατά τμήματα συμφορία τρία τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά δεν είναι τόσο ξεκάθαρο έλεγχος για το δεύτερο τμήμα ηλεκτρονικός έλεγχος Δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. «34 εναντίον, 23 υπέρ, εγκρίνεται, απορρίπτεται μάλλον, το τρίτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται». 467 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 468 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 471 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 473 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 475 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 477 υπέρ 476 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 477 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 52 υπέρ Έλεγχος, θέλετε έλεγχο. 477 ηλεκτρονική επαλήθευση, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 34 με 24 καμία άποχη εγκρίνεται. Συμβαστική 52 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 482 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 486 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 487 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 490 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 489 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 488 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 491 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 492 και 93 και 94 είναι ταυτόσιμες 492 και 493 είναι ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 494 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 495 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 496 υπέρ να ελέγξουμε την 495 ή 494. Έλεγχος της 495. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Πέρας. 22 με 34 απορρίπτατα. 496 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτατα. 497 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 498 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 55 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 56 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 507 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 508 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 57 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Θέλετε να ελέγξουμε. Έλεγχος της 57, συμβιβαστικής 57. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Πέρας. 37 με 20 εγκρίνεται. Πάμε λοιπόν στην 512 και 513 που είναι ταυτόσημες. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 514 υπέρ. κατά δεν είναι ξεκάθαρο ας ελέγξουμε την 514 άρχεται η ψηφοφορία για την 514 πέρας 36-21 ξεκάθαρο αποτέλεσμα εγκρίνεται 5-15 και 5-16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Συμβαστική 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 518 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 519 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 520 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 521 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τώρα πάμε τη λογική σκέψη και τη λογική αναφορές τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Να δούμε τώρα. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 8, 9, 10 και 11 μαζί. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. Συμβαστική 59 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 60 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 61 συμβαστική υπέρ 61 είμαστε τώρα λοιπόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 64 υπέρ έλεγχος για ποια 25 θέλετε να γίνεται επαλήθευση για την 25 ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 25 ξεκινάει πέρας 24 με 32 απερίφθη. Συμβαστική 64 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 29 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 30 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ. κατά απορρίπτεται. Αλλά σηκώνετε το χέρι καλά παρακαλώ. Είμαστε όλοι κουρασμένοι, το καταλαβαίνω. Αν δεν σηκώνετε τα χέρια σας όμως πρέπει να υποθέτω πράγματα για το που πάει η ψηφοφορία. 65 συμβαστική. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 40 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 66 υπέρ κατά, κατά αποχές εγκρίνεται τώρα 46 υπέρ όχι νόμιζα ότι 44 και 45 είχαν καταπέσει. Λάθος. Α, όχι, δίκιο έχετε. Σπαρταρούν και αυτές. 44 και 45 λοιπόν θα τεθούν σε ψηφοφορία από κοινού για την ίδια υπέρ. Κάτα. Αποχές απορρίπτονται. Ας ελέγξουμε, ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά για να είμαστε και σίγουροι. 46 44 μάλλον και 45 ηλεκτρονικά παρακαλώ ψηφίστε. Ελέγχουμε. Ελέγχουμε. Κλοντ με μπερδέψατε. Είδα τον συντονιστή να σηκώνει το, της πολιτικής ομάδας να σηκώνει το χέρι του, άρα όπως πρέπει. Για άλλη μια φορά μια ψήφος παραπάνω στους ελιστές. Διορθώθηκε πέρα της φορείας και γκρίνεται 35 περί 22 κατά. Τώρα, 46 υπέρ. Κατά. Δεν είναι ξεκαθαρό. Μάλλον εγκρίνεται, αλλά δεν ελέγχουμε και ηλεκτρονικά. Σα ζητώ να σηκώνετε ψηλά το χέρι σα. 46. Ψηφίστε ηλεκτρονικά, παρακαλώ. Πέρα φορέ. 30 υπέρ, 26 κατά εγκρίνεται. 47 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίψεται. 49 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 5 είναι απλώς τεχνική, δεν θα τεθεί σε ψηφοφορία. 51 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται και 67 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 56 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 57 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 58 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 59 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 60 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 61 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 62 υπέρ κατά κατά αποχές απορρίπτεται 63 να ελέγξουμε γιατί είναι 62. Να σε ελέγξουμε, ναι. Όλοι κουρασμένοι είμαστε. Σηκώνετε ψηλά τα χέρια σα γιατί συνέχεια ελέγχουμε ηλεκτρονικά και μπερδευόμαστε διαφορετικά. Βλέπω ότι έχει συγκεντρωθεί μια κρίσιμη μάζα από τους συντονιστέ. 62. Παρακαλώ ψηφίστε ηλεκτρονικά. Now, 33 against 20. 33 υπέρ, 23 κατά, εγκρίνεται. 63 υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 64 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 65 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται 66 υπέρ. Κατά. απόχέ, Εγκρίνεται. 68 συμβαστική υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 69 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 72 υπέρ. Κατά. απόχέ. Απορρίπτεται. 73 υπέρ. Κάτα. Αποχές. Εγκρίνεται. 74 υπέρ. Ναι. Νόμιζα ότι εγκρίθηκε 73, αλλά σε ελέγξουμε και ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ 73. Πέρασε τις φορές. ξεκάθαρα απορρίφθηκε. Εβδομήντα τέσσερα. Υπέρ. Κατά. Εάν ούτε οι σοσιαλιστέ δεν μα ξεκαθαρίζουν ποια είναι η θέση του, που είναι δικό σα και ο εισαγητή, τέλο πάντων. Ζητώ συγγνώμη, 74, 74. Ας, ε... Είμαστε ξεκάθαρα τώρα. 74. Πά. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 75 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 76 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται 77. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 78 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 79 υπέρ. Ζητάτε να ελέγξουμε την 78. 78 ηλεκτρονικός έλεγχος. Παρακαλώ ψηφίστε. Πέρας Πέρα Πέρας ψηφορίας είπαμε. 31 υπέρ 26 κατά. Τώρα 79, 79 υπέρ κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 80 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 81 υπέρ. 81 υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε. Δεν ήταν 81 παρακαλώ ψηφίστε ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. «33 έναντι 25 εγκρίνεται, 82 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται». 83 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 84 υπέρ. 84 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 85 υπέρ. Τι θέλετε να ελέγξουμε. Την 83 και την 84 θέλετε να ελέγξουμε. Ωραία. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τροπολογία 83. 83 ψηφίστε παρακαλώ. Και πέρα ψηφοφορίας. Τώρα πέρα ψηφοφορίας. 35 πέρα 23 κατά εγκρίνεται. Και τώρα ξαναθέτω σε ψηφοφορία ηλεκτρονικά την 84 για έλεγχο. Παρακαλώ ψηφίστε. Πέρας ψηφοφορίας. 34 υπέρ 25 κατά εγκρίνεται. 85 υπέρ. Κατά. Οι σοσιαλιστές τι. Υπέρ, υπέρ είμαστε. Μάλιστα, υπέρ είστε. 86, 86 υπέρ. Κατά. Αποχές ε, απορρίπτεται. 87 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 88 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 89 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 90 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 91 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται το 92 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 93 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 94 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 95 υπέρ Εγκρίθηκε, εγκρίθηκε. Διευκρινίζει ο πρόεδρος. Α, ζητώ συγγνώμη, είπα ότι απορρίφθηκε ενώ στην πραγματικότητα εγκρίθηκε με ξεκάθαρη πλειοψηφία. Αλλά σε ελέγξουμε ηλεκτρονικά τώρα γιατί δεν είναι πράγμα αυτό. 94. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. 42 υπέρ, 15 κατά. Ξεκάθαρα λοιπόν εγκρίθηκε. 95 υπέρ, Εδώ πρέπει να ελέγξουμε. 95. Ηλεκτρονική ψηφορία ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας ψηφορία. 28 υπέρ 26 κατά εγκρίνεται. 96 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται.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 και πηγαίνουμε στην τροπολογία 117. 117 υπέρ. Κάτα. Αποχές. Απορρίπτεται. 118 υπέρ. Κάτα. Αποχές. Εκρίθηκε. 119 υπέρ. Κάτα. Αποχές. Εκρίνεται. 120 υπέρ. Κάτα. Αποχές. Εγκρίνεται τελική ψηφοφορία για το σύνολο του κειμένου όπως τροποποιήθηκε, ηλεκτρονικά ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Πέρασε, 33 ψήφοι υπέρ, 7 κατά, 17 αποχές. Συγχαρητήρια, εγκρίθηκε. Ευχαριστούμε κύριε Μωράη. Δεν τελείωσε. Δεν τελείωσε. Έχουμε μια ψηφοφορία ακόμα η οποία δεν είναι απλή. Είναι η αξιολόγηση της δικαιοσύνης στον τομέα των ποινικών θεμάτων και το κράτους δικαίου. Παρακαλώ, πρέπει να ψηφίσουμε ακόμα. Μην λιποτακτείτε άλλη μια ψηφοφορία. Μην εγκαταλείπετε το κλειδονιζόμενο σκάφος, λέει ο πρόεδρος. Please. Please. Παρακαλώ. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ησυχία και συγκέντρωση, παρακαλώ. Τροπολογία 37, υπέρ. Κατά. Αποχές τη Συμβαστική 1, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Γιούρι 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 47. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 48. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 49. Έχει αποσυρθεί 49. 50. Υπέρ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 Εγώ νομίζω ότι εγκρίθηκε, αλλά σε ελέγξουμε. Πέρας <clears throat> για την, το τρίτο τμήμα της συμβαστικής 3. Πέρας. 12.38 απερίφθη. Σύμβαση 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 71 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 69 και 70 που είναι ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές δεκτές. 72 υπέρ κατά αποχές έλεγχος ας ελέγξουμε η ίδια ισορροπία όπως πριν αλλά εκεί πέρα τα μάτια μου με πρόδωσαν δεν είδα πολλά χέρια ας ψηφίσουμε λοιπόν την 69 και την 70 ή συγγνώμη την 72 άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά πέρασε 31-20 εγκρίνεται. Πάμε στην 73. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Γιούρι 5 υπέρ. Έλεγχος για την 73. Άρχεται η ψηφοφορία. 4 με 48. Με τα τσαρούχια περίφθη. Γιούρι 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Γιούρι 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Αιτιολογικές σκέψεις και αναφορές. Τροπολογία 1. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. Γιούρι 1 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Γιούρι 2 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος για τη Γιούρι 2. Γιούρι 2 άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρασε. 21.32. 21-32. Τροπολογία 2 λέει ο πρόεδρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τέσσερα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Έξι. υπέρ. Κατά. Δεν είναι σαφές. Ελέγχουμε την 6. Άρχεται. Πέρας. Είναι θέμα χεριών, λέει ο πρόεδρος. Εγκρίνεται. 7. <clears throat> Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 8. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 9. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 10. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 8. Υπέρ. κατά δεκτή 15 υπέρ κατά δεκτή 16 υπέρ έλεγχος για 15 15 αρχιτη ψηφοφορία πέρας 33-18 εγκρίνεται 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Έλεγχος 16. Άρχεται. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 34-17 εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά όχι Συγκρίνεται. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 29 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή, 30 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται, 31 υπέρ. Έλεγχος για 30. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. 17-34 απορρίπτεται. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 32 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Γιούρι για την αιτιολογική σκέψη ε υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Γιούρι για το F υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 36 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Γιούρι για το C υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Γιούριντι Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Και το σύνολο του κειμένου πως έχει τροποποιηθεί ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Τι έχουμε. Πέρας ψηφοφορίας. 34 υπέρ, 16 κατά, μία αποχή. Κύριε σε νεκρήθη η έκθεσή σας. Συγχαρητήρια. Έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε. Εντάξει, τελειώσαμε για σήμερα. Συνεχίζουμε αύριο τις 9 το πρωί. Σας ευχαριστώ απαξάπαντες. Sorry, Όχι, όχι, όχι. Λυπάμαι. Έχουμε ένα σημείο ακόμα. Πού είναι η συγγήτρια κυρία Γκέντς. Σας παρακαλώ να μείνετε. Για να παρουσιάσει η κυρία Γκέντς το θέμα της δεν θα κρατήσει πολλή ώρα. Κύριε Γκέντς, έχετε το λόγο. Λυπάμαι που σας κρατάω εδώ. Για δύο λεπτά είναι γνωμοδότηση που αποφασίστηκε την τελευταία στιγμή, Πρόεδρος. Παρακαλώ, παρακαλώ, συνάδελφοι εντός εθούσης, συνάδελφοι εντός εθούσης. Σεβασμό, σεβασμό, συνάδελφοι εντός εθούσης, σεβασμό για την εισηγήτρια που έχει το λόγο. Παρακαλώ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τη βοήθειά σας, Πρόεδρε. Η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε ότι θα ήθελε να ετοιμάσει μία έκθεση για τα μαθήματα από το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και επειδή είμαστε στις διαπραγματεύσεις έχουμε τη δυνατότητα να γνωμοδοτήσουμε την τελευταία στιγμή. Έχουμε πίεση χρόνου είναι έκθεση τελευταία στιγμή. Προσπαθούμε να ζητήσουμε συναδέλφου που είχαν εμπλακεί στι διαπραγματεύσει του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου τι θα μα πούν και να συνοψίσουμε τι απόψει του. Αποδεχόμεθα το, ε, τη δουλειά που έκαναν οι συνάδελφοι. Όλοι είπαν ότι ήταν δυσχερέστατε οι διαπραγματεύσει, χωρί να ξέρει κανεί το τελικό, το τελικό ποσό. Πολύ δύσκολο να διαπραγματεύεται κανεί το περιεχόμενο, χωρί να ξέρει ποιο είναι το διαθέσιμο ποσό. Ήταν ε, ήδη δύσκολε πτυχέ που συζητήθηκαν. Επικοδομητικός ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη Προεδρία με τους πόρους για τη δικαιοσύνη όχι με θέματα εσωτερικών. Εκεί υπήρξε συμφωνία λίγο πολύ, σιωπηρή συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Συμβουλίου, μη λαμβάνοντα υπόψη την άποψη του Κοινοβουλίου. Ο διαχωρισμός των πόρων πήρε πολύ χρόνο. Η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ συμμετείχε στην, ε, στον καθορισμό των ποσών, την αξιολόγηση αυτών. Αναφέρονται η κατοξοδότηση ε, πράξεις για τις εφαρμοστικές αποφάσεις δεν το δεχόμαστε διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να ελέγξει έτσι. Ήταν πολύ περιορισμένος ο χρόνος για μας και θέλουμε να αναφέρουμε ότι έχουμε τροπολογία που ζητούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημοσίευσει στοιχεία ώστε η κοινωνία των πολιτών ήδη να μπορεί να χρηματοδοτηθεί και να μην υπάρχει κενό μεταξύ της παλιάς προγραμματικής περίοδου και της νέας, να καλυφθούν οι δαπάνες. Μόνο με τροπολογίες στα αγγλικά μπορούμε να εργαστούμε, διαφορετικά θα μπορέσουμε να τελειώσουμε εγκαίρως. Προθεσμία για τις τροπολογίες το αργότερο πρέπει να είναι 18 Φεβρουαρίου, Φεβρουαρίου επόμενη Τρίτη. Ε, διαφορετικά δεν μπορούμε να επηρεάσουμε εμείς την ψηφοφορία της Επιτροπής Προπολογισμών. Ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Ήθελα να κάνω ό,τι μπορώ και να συμπεριλάβω στο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία στην ε, έκθεση. Μιλάει ένα συνάδελφος, λέει ο πρόεδρος. Σας παρακαλώ λοιπόν, μην κάνετε φασαρία. Συγκέντρωση θέλω παρακαλώ. Δεν φαίνεται τόσο ενδιαφέρον το θέμα όσο η NSA και το θέμα του κράτους δικαίου κλπ. Αλλά είχα την ευκαιρία να πω τι μάθαμε από τις διαπραγματευτικές διαδικασίες για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Δεν πετύχαμε συμπληρωματικούς πόρους, άρα δεν τους ενδιαφέρω. Ευχαριστώ για τη συνεισφορά σας. Προσπάθησαμε να λάβουμε υπόψη τις απόψεις των διαπραγματευτών και λυπούμεθα, αλλά δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να μπορέσουμε να επηρεάσουμε την κατάσταση παρά να βάλουμε προθεσμία 18 Φεβρουαρίου την επόμενη Τρίτη και τα έγραφα στα αγγλικά. Ζητώ συγγνώμη. Ευχαριστώ για την παρουσίασή σας για το παρουσίαση του σχεδίου εκθέσεως για, το, για τα θέματα που αφορούν το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Δεν ξέρω αν κάποιος θέλει να πει κάτι, αν κάποιος έχει να σχολιάσει. Θέλετε να πείτε κάτι. Ναι, βεβαίως, κύριε Μαρινέσκου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ καλή αυτή η έκθεση. Η γνωμοδότηση πρέπει να αναφέρουμε κάποια γενικά πράγματα διότι στη διαπραγμάτευση του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου έμεινε εκτός το Κοινοβούλιο κατά την άποψή μου. Τα ποσά αποφασίστηκαν στο Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και είμαστε υποχρεωμένοι να πούμε ναι ή όχι. Αυτός είναι ο κανόνας. Όμως μπορούμε να κάνουμε περισσότερα αν προσεγγίσουμε κάθε κεφάλαιο, κάθε ευρωπαϊκή πολιτική μέσω συναποφάσεως, διότι εκεί έχουμε εξουσία. Συμπεριλαμβανομένων και των ζητημάτων εσωτερικών, να δημιουργήσουμε κάτωθεν τον προϋπολογισμό και ουχή άνωθεν. Αυτή είναι η κανονική μέθοδος καταρτήσεως του προϋπολογισμού. Να μην προσπαθήσουμε να επιβάλλουμε ευχολόγια περίπλοκα αλλά να προβούμε σε ανάλυση, να λύσουμε όλες τις ευρωπαϊκές πολιτικές και τι απαιτείται για να πετύχουν τους στόχους τους οι πολιτικές. Αυτή είναι η συνεισφορά μου, αν επιτρέπετε την εκφράσω. Συμφωνείτε κυρία Γκάντς, λέει ο Πρόεδρος. Βεβαίως, βεβαίως. Βλέπω και την κυρία Λάμπερτ που κάτι θέλει να πει. Με τα χαράς να το σκεφτώ αυτό. Αλλά να μιλήσει η κυρία Λάμπερτ. Η κυρία Λάμπερτ και για την ομάδα μας πρέπει να πω ότι συμφωνούμε με την κατεύθυνση που ακολουθεί η γνωμοδότηση. Έχουμε μία-δύο τροπολογίες που θα θέλαμε να υποβάλουμε για κάποιες διαπραγματευτικές θέσεις, αλλά αυτό που αναφέρθηκε για την έλλειψη συμμετοχής του Κοινοβουλίου, όπως τα επιθυμούσαμε, ή θα έπρεπε να γίνει, έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι κάτι το οποίο όσον αφορά τον εσωτερικό συντονισμό του Κοινοβουλίου πρέπει να εξεταστεί την επόμενη φορά. Διότι το Κοινοβούλιο δεν είχε συντονισμένη θέση σε κάποιες φάσεις και αυτό δεν βοήθησε. Η κυρία Γκέντς, δύο λόγια να πω, δύο φράσεις. Υπάρχει προθεσμία πολύ κοντινή και λυπάμαι με τα χαράς να λάβω τις τροπολογίες σας της, του κυρίου Μαρινέσκου και της Τζέιν Λάμπερτ. Δεν με ενδιαφέρει η κριτική, δεν με ενοχλεί. Μπορούμε να το στείλουμε αυτό το έγγραφο σαν τροφοδότη του προβληματισμού της Επιτροπής Προϋπολογισμών, που και αυτή είναι στριμωγμένη χρονικά. Θέλουμε να είμαστε θετικοί όσον αφορά κάποιες πτυχές, κυρίως όσον αφορά τα δικά μας θέματα, όχι τα θέματα εσωτερικών, Εκεί ήταν δυσχερέστατη η κατάσταση και δεν ελήφθησαν υπόψη οι απόψεις του Κοινοβουλίου. Είμαστε πιο κριτικοί με τα χαράς να συμπεριλάβω τις ε, τροπολογίες σας. Προθεσμία είναι 18 του Φεβρουαρίου, Τρίτη. Δύο εργάσιμες μέρες ακόμα. Δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε αλλιώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ για την παρουσίαση. Την παρουσίαση που κάνατε τα καταφέραμε. Ξεπερδέψαμε γρήγορα αρκετά για σήμερα. Θα τα πούμε αύριο στις 9 το πρωί. Σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ.